και τους σοσιαλιστούς αιτήματα για αλλαγή στη σύνθεση επιτροπών και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις,